All right. Please, colleagues, take your seats. The vote is a... Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι γιατί αρχίζει η ψηφοφορία. Now the first vote is a roll call vote. Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει με ονομαστική κλίση, γι' αυτό παρακαλώ τοποθετήστε τις κάρτες σας στο μηχάνημα.